από 70 χρόνια στις 17 Ιανουαρίου του 1945 απελευθερώθηκε από τους Σοβιετικούς στρατιώτες, του Σοβιετικό στρατό, το στρατόπεδο του Auschwitz. Οι πρώτες εικόνες που αντίκρισαν οι στρατιώτες αυτοί συγκλονίζουν ακόμη και μέχρι σήμερα τον κόσμο. Βουνά από πτώματα, κρεματόρια, βουνά από παπούτσια γυαλιά, μαλλιά ανθρώπων, συντρίμια λαιλατημένων ζώων. Μαρτυρούσαν περισσότερο το θάνατο οι εικόνες αυτές παρά τη ζωή. Οι εικόνες αυτές έχουν χαραχθεί ανεξίτηλα στη συλλογική μνήμη του ανθρώπου. Για τους περισσότερους από τους κρατούμενους στο Auschwitz η σωτηρία έφτασε με μεγάλη καθυστέρηση. Πάνω από ένα εκατομμύριο άνθρωποι δολοφονήθηκαν σε αυτό το στρατόπεδο της εξολόθρευσης, της εξόντωσης, από το πείνα, της ασθένεια, από εγκληματικού χαρακτήρα ιατρικές ε, δοκιμές και πάνω απ' όλα από το τη συστηματική θανάτωση στα... στους θαλάμους αερίων από την Ολλανδία, τη Γαλλία, την Πολωνία, την Ελλάδα, άνθρωποι κάθε πίστης από όλη την Ευρώπη, Συντή και Ρωμά, άνθρωποι με αναπηρίες, άνθρωποι ασθενείς, ομοφιλόφιλοι, πολιτικοί κρατούμενοι, εχμάλωτοι πολέμου και πάνω απ' όλα αμέτρητα παιδιά. Αυτό το οποίο συγκλώνησε τον κάθε επισκέπτη του Auschwitz έκτοτε. Αμέτρητα παιδιά. Αυτούς τους οποίους είχαν χαρακτηρίσει με την απάνθρωπη ιδεολογία των Ναζί ως υπανθρώπους, για τους οποίους η ανθρώπινη ζωή δεν είχε καμία αξία. Αυτοί οι άνθρωποι θέλησαν να εκριζώσουν αυτή τη ζωή, αυτές τις ζωές. Το Auschwitz δεν ήταν ο μόνος, αλλά ο κεντρικός τόπος του μαζικής εξόντωσης για την ιστορία του ανθρώπου αυτών των ζώων. Αυτός ο τόπος παραμένει μία φωνή αγωνίας, μια φωνή προειδοποίησης για όλη την ανθρωπότητα με αυτή την ιστορία που έχει γραφτεί στα στρατόπεδα εξόντωσης. Μια φωνή απελπισίας, μια φωνή προειδοποίησης. Αυτό είναι το Auschwitz και όλα τα στρατόπεδα. Μπορεί την προσωπική ποινική ευθύνη να την πήρε ο κάθε ένας από τους ε, υπετίους μαζί του στον τάφο. Αλλά η συλλογική ευθύνη ανήκει σε όλους μας και πάνω απ' όλα στο λαό στον οποίο ανήκω εγώ το γερμανικό η ευθύνη ποτέ να μην επιτρέψουμε να ξανασυμβούν αυτά τα πράγματα. Είναι μια ευθύνη που ανήκει σε εμά τις επόμενες γενναίες στον αιώνα των αιώνων. Ε, η ιστορία μπορεί να μην επαναλαμβάνεται. Αλλά ο τρόπος με τον οποίο προχωρούμε, με τον οποίο βλέπουμε τόσο την ιστορία μας όσο και το παρόν μας, είναι ο τρόπος με τον, στον οποίο εμείς έχουμε την ευθύνη. Και γι' αυτό πρέπει να θυμόμαστε ότι συνέβη το αδιανόητο στο Auschwitz. Και γι' αυτό πρέπει κάθε μέρα να αγωνιζόμαστε για την ελευθερία, για την αδιαπραγμάτευτη αξιοπρέπεια του ανθρώπου. Γι' αυτό κάθε μέρα πρέπει να αγωνιζόμαστε ενάντια στην επάνωδο ιδεολογιών και κοσμοθεωριών οι οποίες στηρίζονται στο μίσος, την ξενοφοβία, τον αντισημιτισμό, τον ακραίο εθνικισμό, την αδιαλαξία. Γιατί σήμερα, 70 χρόνια μετά την απελευθέρωση του Auschwitz, υπάρχουν ακόμα Εβραίοι στην Ευρώπη που φοβούνται για την ασφάλεια τους και φοβούνται ότι μπορεί να χάσουν τη ζωή τους. Αυτό πρέπει να μας συνταράξει. Σήμερα πρέπει να σταθούμε όλοι μαζί δίπλα τους, απέναντι στο φόβο και να μην επιτρέψουμε να επιμολυνθούμε από το μίσος, αυτό το οποίο κίνησε το χέρι των δολοφόνων στο Παρίσι. Πρέπει να δώσουμε την απάντησή μας αποφασιστικά και να πούμε ότι δεν θα απαντήσουμε στη βία με νέα βία, αλλά ότι θα αγωνιστούμε για τις αξίες και την αξιοπρέπεια του κάθε ενός ανθρώπου και θα την προστατέψουμε. Αυτό είναι το καθήκον που έχουμε σήμερα, 70 χρόνια μετά το τέλος του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου και την απελευθέρωση του Auschwitz. Εδώ, στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο που αποτελεί και την έκφραση τη συνέλευση των λαών της Ευρώπης, μια πολυεθνική συνέλευση, οφείλουμε εμείς να αναλάβουμε το πρώτο βήμα. Ευχαριστώ. Επόμενο θέμα στην ημερήσια διάταξη. Δήλωση του Συμβουλίου και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής απολογισμός της Ιταλικής Προεδρίας. Και έτσι καλωσορίζω τον Πρωθυπουργό της Ιταλίας, κύριο Ρέντσι. Έχετε το λόγο παρακαλώ.